Nous Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Συγγνώμη να ζητήσω, γιατί περιμένατε στο διάδρομο μέχρι να αρχίσουμε. Επόδεινο. Συγγνώμη, αλλά άργησε η συνεδρίαση των συντονιστών, γιατί έχουμε δύσκολα θέματα να συζητήσουμε. Θα περάσουμε τώρα στο ζήτημα της ε, συνένεσης επί της ανθρωπιστικής βοήθειας θα κάνουμε έναν απολογισμό και θα παρουσιαστεί η εκτέλεση του σχεδίου, του σχεδίου δράσης. Ο κύριος Τρίφλερ θα πάρει πρώτα το λόγο, ο οποίος ε, θα ξεκινήσει την ε, συζήτηση και θα ε, παρουσιάσει τους υπόλοιπους ομιλητές. Voilà. Donc, euh, στις 18 Δεκεμβρίου 2007 οι, πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου υπέγραψαν τη συνένεση επί της ανθρωπιστικής βοήθειας με σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συνεργαστεί για την εκτέλεση του σχεδίου δράση ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό στι διαπραγματεύσει ε, σε ένα πιο δύσκολο ανθρωπιστικό πλαίσιο. Η συνένεση είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τη βοήθεια ε, την ανθρωπιστική γιατί εξασφαλίζει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα κοινό όραμα, όπως επίσης και μια συγκεκριμένη στρατηγική που μπορεί να βοηθήσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πλήττονται από τις συγκρούσεις και από τις φυσικές καταστροφές και επομένως ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει υπέρ ε, των ε, αξιών ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν. Το 2008 ε, υπήρξε ένα σχέδιο δράσης ε, με συγκεκριμένα μέτρα εκτέλεσης ε, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων που προορίζονται για τους δωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διευκολύνουν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Για να μπορέσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια Βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ερυθρά μισέλινο και στον Ερυθρό Σταυρό και στη, στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ σαφή τρόπο τονίζει τη σημασία του πλουραλισμού αυτού των εταίρων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλέσαμε στη συζήτηση τον Αντουάν Ναζερά Ρασέλ από το ΕΚΟ, ε, η κυρία, ε, την κυρία Ζενεβιέβ ε, Ρες από την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει το 2009 μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της εφαρμογής της συνένεσης στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των εταίρων της. Ε, είναι εδώ και ο κύριος Πίτερ Ζάγκλ, ο Γενικός Διευθυντής ε, της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας ως εισηγήτρια για την ανθρωπιστική βοήθεια θα καταρτήσω, θα συντάξω ένα κείμενο σε σχέση με την εφαρμογή της ε, συνένεσης ανθρωπιστικής βοήθειας που θα ψηφίσουμε το φθινόπωρο. Πρέπει να συζητήσουμε και τις επιτυχίες ε, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις στο πλαίσιο της ε, συνένεσης ανθρωπιστικής βοήθειας και του σχεδίου δράσης και ελπίζω να ε, γίνει η συζήτηση, να συνεχιστεί η συζήτηση στην ομάδα εργασίας ε της ευρωπαϊκή Επιτροπής, ε, καλώντας εκπροσώπους ε, της συνένεσης αυτής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Ο κύριος ε, Πίτερ Τζάγκλ έχει το λόγο για 7 λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Στρικέ που μας ξεκαθάρισε τα πιο σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την ε, συνένεση και επιπρόσθετα για το τι μας ε, περιμένει σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσης που συνοδεύει την Ευρωπαϊκή Συνένεση. Ε, ήρθε η Επιτροπός χτες εδώ στην Επιτροπή σας ε, και γι' αυτό το πολύ σημαντικό πολιτικό έγγραφο που εγκρίθηκε από τα τρία όργανα. Νομίζω ότι δόθηκε το πιο σημαντικό μήνυμα χθε ότι μέχρι σήμερα μας έχει εξυπηρετήσει πολύ καλά η συνένεση και ε, θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Έτσι λοιπόν θέλουμε να κινηθούμε φιλόδοξα και ε, να θέσουμε ξεκάθαρους στόχους και δεσμεύσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνένεση αυτή είναι τόσο σκόπιμη με σήμερα όσο ήταν και το 2007 γιατί παρουσιάζει κύριες προσκλήσεις για το πώς ε, θα διασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα στην απάντηση ε, που δίνουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, πώς θα υπάρχει καλό συντονισμός και αλληλεπίδραση. Υπογραμμίζει το ευρωπαϊκό όραμα εταιρική σχέσης στην ανθρωπιστική δράση, αναγνωρίζοντας ε, την αξία της ποικιλομορφία ε, στην ανθρωπιστική εταιρική σχέση και συμπεριλαμβάνουμε εκεί και συγκεκριμένου ρόλους ε, για τον ΟΗΕ, για τον ε, Ερυθρό Σταυρό και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται στον ανθρωπιστικό τομέα και φυσικά διασφαλίζουμε και το γενικό συντονιστικό ρόλο της ΟΤΣΑ εμείς ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε αποκτήσει θεσμικό βάρος ε, και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε το όργανο που μας ε, βοήθησε στο έργο μας και προστίθεται τώρα στο ε, τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας γιατί έχουμε φυσικά τώρα όπως γνωρίζετε και μία επίτροπο για την ανθρωπιστική βοήθεια ε, και ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ε, Κομισιόν παρουσιάζει πάρα πολύ υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά ε, την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς εργαστήκαμε πολύ σκληρά για την οθέτηση αυτών των προτύπων και ουσιαστικά εμείς προωθήσαμε το θέμα της στρατηγικής ανάλυσης και της ανταλλαγή πληροφοριών και άλλων θεμάτων. Όμως, δυστυχώ. Ε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έχουμε επιτυχεί μέχρι τώρα, καθώς μπήκαμε σε ένα έτος ε, που είχαμε τον καταστροφικό σεισμό στην ε, ΑΙΤ και πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο δραματικό γεγονός. Ε, μία από τις πιο ευάλωτες χώρες ε, της Αμερικής χτυπήθηκε. Και να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 11 Ιανουαρίου η ΑΕΤ ήταν ε, ήδη ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μας, όμως υπό την κατηγορία ξεχασμένων κρίσεων και τώρα ίσως πρέπει να βγει από την κατηγορία αυτή μετά από το σεισμό του Ιανουαρίου υπήρξε συνένεση για την ε, διεθνή υποστήριξη που πρέπει να δοθεί, όμως ε, θέλουμε αυτή η συνένεση να γίνει περισσότερο γνωστή. Πρέπει ε, ουσιαστικά η κοινότητα να λάβει πιο σημαντικό ρόλο και αυτό να συμπεριλάβουμε πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στους δωρητές. Επίσης, πρέπει να ε, απευθυνθούμε περισσότερο στα Εθνικά Κοινοβούλια και θέλουμε την υποστήριξή σας για να το πετύχουμε αυτό αποτελεσματικά, όπως ε, θέλουμε και να συζητήσουμε και με άλλους πρωταγωνιστές ε, που ανέφερε χθε η Επίτροπος, όπως είναι η πολιτική και η στρατιωτική. Μάλλον Πρώτα με του πολιτικούς θα πρέπει να μιλήσουμε για κατόπιν με του στρατιωτικού. όμως ε, και οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να συμμετέχουν στι συζητήσεις μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η απάντηση στην κρίση, η αποκρίση στην κρίση ε, ε, θα δίνεται όταν χρειάζεται και πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να εξηγούμε γιατί ε, δεσμεύουμε κάποια κονδύλια για συγκεκριμένους σκοπούς ε, και όχι για κάποιο άλλους. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση η οικοδομή ικανότητες πολιτικής προστασίας, εμπειρογνωμοσύνη που χρησιμοποιούνται σωστά και με ένα συμπληρωματικό τρόπο. Αυτό αποτελεί τη ρεχοκοκαλιά της ενδιάμεσης αναθεώρησης του σχεδίου δράσης η Κομισιόν ξεκινά αρχικά τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη γιατί θέλει να ακούσει τι ανησυχίε των υπόνων. Εμεί θεωρούμε ότι η αναθεώρηση αυτή είναι η κυρία ευκαιρία για να παγιώσουμε την όθηση και την υποστήριξη πίσω από τη συνένεση και να επικεντρωθούμε σε κάποιε κυρίε προτεραιότητε. Βασικά, θέλουμε η διαδικασία τη ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράση να είναι όσο το δυνατό πιο ανοιχτή και συμμετοχική, όπω ήταν η διαδικασία που οδήγησε στην ίδια τη συνένεση. Και στο πνεύμα αυτό ήρθα εδώ σήμερα το πρωί ενώπιόν και φυσικά ε, ευχαρίστως ε, να ακούσω τα σχόλιά σας και αν έχετε και ερωτήσεις με στη σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Αντουάν Ζεράρ από την ΩΣΑ για 7 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκλησή σας, αλλά και για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος την ε, όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ανθρωπιστικά ζητήματα υπό την ηγεσία βέβαια ε, αρμόδιας εισηγήτριας. Είμαστε, όπως υπόθηκε, σε μια κρίσιμη χρονιά σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή της συνένεσης αυτής. Όπως ε, είπε ο Τζον Χόλμς από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 29 Ιανουαρίου 2008 η συνένεση σημαίνει σοβαρή δέσμευση για την αρχή της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και όπως ε, υπόθηκε ήδη και από τον Πίτερ, η ανταπόκριση στις ανάγκες που υπάρχουν ε, είναι πολύ σημαντική και ειδικότερα βάσει της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας, ε, ε, είναι αρχές και αυτές που πρέπει να ακολουθούν. Και στον ΟΗΕ αποτελεί ζήτημα προτεραιότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας ο κεντρικός συντονιστικός λόγος, ρόλος της υπηρεσίας για, την ανθρωπιστική βοήθεια, της ΟΤΣΑ, έχει να κάνει με συγκεκριμένα άρθρα της ε, συνένεσης και αν μου επιτρέπετε θα σας ε, εξηγήσω πώς μπορούν ε, πρακτικώς να εφαρμοστούν. Αναφέρομαι λοιπόν στο άρθρο 25. Επίσης χαιρετίζουμε την πλήρη έγκριση της μεταρρύθμισης ανθρωπιστικής βοήθειας και ειδικότερα την αναφορά σε ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 67. Επίσης η αναγνώριση των ε, κατευθυντηρίων ε, για τη χρήση ε, πολιτικών και στρατιωτικών μέσων, τη χαιρετίζουμε μεν, και η αντίδρασή μας ε, στην κατάσταση στην ΑΕΤ έδειξε πόσο σημαντικό είναι η δράση μας να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές ε, της, ε, του Όσλο και πώς αυτό το ζήτημα πρέπει να είναι στο πλαίσιο ε, της δουλειάς του συντονιστή ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας και είναι κάτι το οποίο, του οποίο επικεφαλής ε, πρέπει να είναι η ε, κοινότητα των πολιτών, η κοινωνία των πολιτών. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Δώστε μου τη δυνατότητα να αναφερθώ στο άρθρο 15, το οποίο αναφέρει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εργαλείο διαχείρισης της κρίσης. Ε, χαιρετίζουμε το σχέδιο δράσης ε, την έγκριση δύο δράσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αναθεώρησή του. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω μεγαλύτερη δέσμευση από πλευρά ε, των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή υπάρχουν θεσμικέ αλλαγέ λόγω τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει μεγαλύτερη εξουσία ε, και για τα ζητήματα τη νομοθεσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά τα ανθρωπιστικά, λοιπόν, θα μπορούσε το, το, το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ε, να είναι επικεφαλής μιας τέτοιας προσπάθειας με γνώμονα τις αρχές. Πέρα από, την, από τα πολιτικά ζητήματα επίσης μπορείτε να ενθαρρύνετε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα να εφαρμόσουν ε, τις, την καλή πρακτική ε, των δωρητών όπως αναφέρεται στο άρθρο 96. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ορισμένους πρακτικούς τρόπους για να προχωρήσουμε για το θέμα της συνένεσης, εκτός από την αναθεώρηση και την έκθεσή σας ε, που περιμένουμε εναγωνίως να συνεισφέρουμε σε αυτήν. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαίνει ότι θα έπρεπε να πρωτοστατήσει σε σχέση με την εφαρμογή της συνένεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων ε, και σε ευρύτερο σημείο, πέρα, σε ευρύτερο πλαίσιο ε, στις δικές σας ε, περιφέρειες, ε, στο πλαίσιο των εθνικών κυβερνήσεων ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική συνέλευση που υφίσταται, η συνεισφορά θα είναι θέμενη αξία. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που παρατήρησα στις τακτικές επαφές μου με το Κοινοβούλιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ, 21 χώρες ε, του ΝΑΤΟ θα είχαν υπογράψει ε, την ε, συνένεση αυτή αν είχαν γνωρίσει καλά σε τι συνίσταται. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και να συμφωνήσω σε αυτό το σημείο με τον Πίτερ ότι η συνένεση πρέπει να είναι ένα εργαλείο όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και στις πρωτεύουσές σας. Υπάρχει λοιπόν η ανθρωπιστική υπηρεσία και εμείς ως συντονιστές με μεγάλη χαρά θα συμβάλλουμε στις υποστηρίξεις του στην υποστήριξη των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό χαιρετίζουμε ιδιαίτερα ε, την πρωτοβουλία αυτή για μεγαλύτερες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ομάδας Ε. ε Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατρίν Σιπτ έχει το λόγο τώρα από το Voice για 7 λεπτά. Καλημέρα σας. Εγώ εκπροσωπώ τις 87 ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που απασχολούνται στον ανθρωπιστικό τομέα ως Πάμε σε the και τα λοιπά και χαίρομαι ε, που εδώ έρχομαι σε ε, επαφή με το νέο κοινοβούλιο καθώς οι οργανώσεις μας έχουν δεσμευτεί πάρα πολύ ε, και έχουν συμμετάσχει ενεργά στο θέμα της συνένεσης. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό που συμπληρώνει οι και ισχυροποιεί και τη θέση μας ε, διεθνώς. Χαιρόμαστε που μας καλέσατε εδώ σήμερα και θέλουμε να απευθυνθούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απευθύνουμε έκκληση να δεσμευτεί για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ε, της συνένεση τόσο όσο και το παλιό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή αρχή. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε καταρχήν να καλωσορίσουμε. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τη ΓΔΕ όταν αναπτύξαν ε, τι ε, διάφορε κατευθυντήριε γραμμέ για τη χάραξη πολιτική ε, και υπήρξε πολύ στενή συνεργασία με τις ΜΚΟ. Το εκτιμούμε αυτό και εμεί θεωρούμε ότι είναι ευπρόσδεκτη εμπειρία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται πάρα πολλά χρόνια στον τομέα. Είναι όμω δύσκολο να δούμε πώ τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει τη συνένεση. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως ανέφερε ε, και ο κ. Ζεράρ, ε, νομίζω ότι η Προεδρία ε, πρέπει να αναφέρει πώς τελικά συνολικά αλλά και μεμονωμένα τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει το σχέδιο δράσης και τη συνένεση μέχρι τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω διάλογο. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο θέμα του διαλόγου για ανθρωπιστικά ζητήματα που αναφέρθηκαν και από την Επίτροπο χθε. Αυτά ε, μας ανησυχούν πάρα πολύ σε σχέση με τις, την κατάσταση στην οποία εργάζονται ε, οι άνθρωποι επιτόπου, ε, οι αρμόδιοι για την παροχή βοήθειας. Ξέρω ότι αυτό απασχολεί και τη σημερινή Επίτροπο και νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και ε, σε επίπεδο θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει πολλά να γίνουν. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες. Ε, πρέπει να καταλάβει ο καθένας ε, την εντολή και το ρόλο του άλλου και νομίζω ότι ε, από την πρόσφατη κατάσταση στην ΑΕΤ κατέστη σαφέ ότι καταρχήν χρειαζόμαστε ένα σαφή προσδιορισμό της εντολής και των ρόλων των διάφορων πρωταγωνιστών ε, στην ανθρωπιστική κρίση των διάφορων συμμετεχόντων. Αυτή είναι πραγματική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο ε, σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές πληροφοριών ε, με την Επίτροπο αλλά και την πρόθεση των θεμάτων αυτών. Ένα άλλο θέμα είναι η πολιτική προστασία. Θεωρώ ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος, ε, ως προς τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διάφορων μηχανισμών ε, της Ένωσης, έτσι ώστε η πολιτική προστασία να είναι και τώρα στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΟ. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση ως προς την εφαρμογή και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ε, προκειμένου να το θέσουμε σε εφαρμογή, αλλά νομίζω ότι ήδη το πρώτο βήμα, δηλαδή να κάνουμε μια αξιολόγηση των κοινών αναγκών επιτόπου, είναι σωτικό και πρέπει να δυσφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, συγγνώμη, ότι η πολιτική προστασία συμπληρώνει την ανθρωπιστική, ότι καλύπτει τα κενά που η παραδοσιακή πρωταγωνιστές δεν μπορούν να καλύψουν, αλλά αυτό γίνεται με στενή συνεργασία και συντονισμό. Και φυσικά είναι πρόκληση να δούμε πώς μπορούμε να τελοποιήσουμε αυτά στο το δυνατό καλύτερα ένα άλλο θέμα ε, που μας απασχόλησε. Η συνένεση μιλά για τις αρχές της ε, εταιρική σχέσης, αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ του ΙΕΤΣ, οικογένεια του Ερθρού Σταυρού και των ΜΚΟ. Έχουμε μια παγκόσμια ανθρωπιστική πλατφόρμα η οποία έχει εγκρίνει αυτές τις αρχές εταιρικές σχέσεις και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη εδώ μπορούν να διαδραματίσουν ε, κάποιο ρόλο μέσω των επιτροπών ε, στις, ε, ε, στους οργανισμούς του ΙΕ για να προωθήσουν τις αρχές της εταιρική σχέσης, γιατί η εταιρική σχέση αποτελεί ένα κυρίο χαρακτηριστικό μεταξύ κρατών, μελών, μη καπαόμικρων, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Πρέπει να προωθηθεί λοιπόν αυτό. Το τρίτο θέμα συνίσταται περισσότερο στη συμπληρωματικότητα των διαφορών μηχανισμών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή τη ε, παρά στην ολοκλήρωση. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επαγρυπνεί το Κοινοβούλιο και να το παρακολουθεί αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να προβάλλουμε τι ανθρωπιστικέ προσπάθειε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την καλή δουλειά που γίνεται μέσω από τι ΜΚΟ των Ερυθρό και τους οργανισμούς του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε κατά κάποιο τρόπο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να βασίζεται στις ανθρωπιστικές αρχές ε, της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με όλους τους υφιστόμενους μηχανισμούς. Ε, που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτή είναι μια πρόκληση που όλοι πρέπει ε, να έχουμε κατά νου. Και το τελευταίο μου σημείο αφορά την ε, λογοδοσία ή συνένεση. Εστιάζει ιδιαίτερα στο θέμα της λογοδοσίας όχι μόνο από τις ΜΚΑ μικρών προς τους δωρητές, αλλά και από τους δωρητές και τις ΜΚΑ μικρών και από άλλους πρωταγωνιστές και συμμετέχοντες προς ε, τα άτομα που, είναι παραλήπτες της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση και πρέπει να δεσμευτούμε όλοι σε αυτό ότι ε, και τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δωρητέ ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, το έγγραφο τη συνένεση για μα είναι έγγραφο αναφορά. Πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα στο μέλλον με την αρχιτεκτονική που έχουμε τώρα στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς ε, είναι πιο ενδυναμωμένος τώρα ο τομέα. και επίσης ε, πρέπει να επανερχόμαστε στο έγγραφο αυτό, να, λέμε, να δούμε για τα συγκεκριμένα θέματα τι λέει το έγγραφο τη συνένεση. Κάτι ακόμα, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη διαβούλευσης των ΜΚΟ, κυρίως σε ε, ό,τι αφορά και ε, την ΕΚΟ, αλλά φυσικά τη διαβούλευση και με τα Ηνωμένα Έθνη και με τον ε, Ερυθρό Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας ζητάνε τις συμβουλές μας, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η ποιότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της συνένεση είναι κάτι που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο ανθρωπιστική εκούσια βοήθεια και αυτό υποτίθεται θα ξεκινήσει το 2011 και εμεί φυσικά θέλουμε να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώ μπορεί να γίνει όσο δυνατόν καλύτερη εφαρμογή. Σα ευχαριστώ πολύ και ανυπομονώ για περαιτέρα διάλογο μαζί σα για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα και σα ευχαριστώ για τη δεσμευσή σα. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ζενεβιέβ του ΣΕΑ από την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για πέντε λεπτά. Σήμερα, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρου τη Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού είναι μεγάλη χαρά για μένα να συμμετέχω στη σημερινή ε, ακρόαση που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Αυτοπιστική Βοήθεια, που είναι ένα έγγραφο πάρα πολύ ε, χρήσιμο. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, ε, ότι η Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό ε, στι διαπραγματεύσει και την επεξεργασία της συνένεσης, σύμφωνα με την εντολή που είναι να προστατεύει τα θύματα εσωτερική βία και ενόπλων σειράξεων με ανεξάρτητο τρόπο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ευρωπαϊκά όργανα και ειδικότερα τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την εμπιστοσύνη της. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι εμείς θέλαμε την ε, εμπειρία μας, τη μεθοδολογική και την επιχειρησιακή να την ε, μεταλαμπαδεύσουμε ειδικότερα στο πλαίσιο το διεθνές, ε, στην, στο πλαίσιο της των τομεακών πολιτικών, ε, όπως για παράδειγμα στην ε, ενίσχυση των τοπικών ε, δυνατοτήτων στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι προτάσεις μας σε γενικές γραμμές ελήφθησαν υπόψη και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει και όσον αφορά τις μελλοντικέ προκλήσεις για την εφαρμογή της συνένεσης, του σχεδίου δράσης. Ε, πρώτον, ε, το διεθνές δίκαιο, η διάδοσή του, ε, η εταιρική σχέση και ο συντονισμός και επίσης η βοήθεια στο πλαίσιο της μετάβασης. Όσον αφορά την προώθηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες που ελήφθηκαν το 2009 από την Τσεχική και την Σουηδική Προεδρία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ε, την προώθηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για το διάλογο με τις τρίτες χώρες ε, για το ζήτημα αυτό. Η Επιτροπή μας ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά όργανα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να εφαρμόσει την απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2008 όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσον αφορά τη συνεισφορά μας και της Διεθνούς, ε, και της διεθνούς Ομοσπονδίας Ρυθρού Σταυρού, τον Ιούνιο του 2009 με την επέτειο της μάχης του Σολφερίνο διακηρύξαμε και πάλι ε, την σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο των θεμελιωδών ε, αρχών μας, που για μας ε, είναι και επιχειρησιακά μέσα που μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Σήμερα η πρόκλησή μας είναι να μην χρησιμοποιούνται με στρεβλό τρόπο οι αρχές αυτές ε, από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Και για να ολοκληρώσω για το πρώτο αυτό ζήτημα, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων ε, για, την, ε, για το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο, είμαστε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να ζητήσουμε να μας λάβετε υπόψη, να σας πούμε επίσης ότι είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεστε. Όσον αφορά τώρα το συντονισμό και τη συνεργασία, στις χώρες όπου δραστηριοποιούμεθα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην διάδραση της στρατηγική με την Ερυθρά Ημισέλινο και γι' αυτό ακριβώς με στοχευμένο τρόπο υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας ε, για την ενίσχυσή του. Το 2010 θα συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με ε, χώρες όπως το Αφγανιστάν, ε, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Σομαλία, η Εμένη και ο κατάλογος είναι μακρύς για μας ε, η μεγάλη πρόκληση είναι να ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση και να έχουμε την υποστήριξη των δοητών. Όσον αφορά τώρα το συντονισμό και τη συνεργασία με τους άλλους εταίρους μας, έχουμε πολύ στενές επαφές, ε, στενές επαφές επιτόπου και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και με τις, ε, τους, τα, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και όσον αφορά τώρα την ανταπόκριση στις ανάγκες ε, κοινωνιών που βρίσκονται σε μετάβαση, Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ καλά, να ενισχύσουμε ε, την κοινωνία των ε, πολιτών και την προώθηση της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να φτάσει αυτή στις πιο ευάλωτες ομάδες για ζητήματα όπως η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη κλπ. Όσον αφορά την επιτόπου υποστήριξή μας, ε, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθήσουμε να προωθούμε μια καλύτερη γνώση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ως ε, επιχειρησιακού εργαλείου που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα οι, ανθρω... οι ανθρωπιστικής ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου, ενισχύοντας τις τοπικές κοινότητες ε, και ε, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ανθρωπιστικές οργανώσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ε, επαφιέμεθα στην υποστήριξή σας ε, και για το σχέδιο δράσης αλλά και για την αναθεώρηση και ελπίζουμε το έγγραφο αυτό να γίνει ευρέως γνωστό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κρόνεμπερκ από τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η Διεθνής Ομοσπονδία και η ενώσει του ε, Ερυθρού Σταυρού θεωρούν ότι αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ καλό και καθορίζει σαφώς τις αρχές της ε, ανθρωπιστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε την ευκαιρία που έχουμε να συμβάλλουμε στην ε, διαδικασία διαβούλευσης που οδηγεί στην έγκριση του συμβιβασμού για το πρόγραμμα δράσης. Η Διεθνή Ομοσπονδία καλωσορίζει τις, τις, τα επιτεύγματα όπως η δημιουργία της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου που είπε ο κύριος Άγκολίδη, και τον ορισμό των διαφόρων ε, κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές που έγιναν από κοινού με, τους, ε, με την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Θεωρούμε όμως ότι ακόμη υπάρχει ε, πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και σε επίπεδο των μελών για να επιτευχθούν οι υποχρεώσεις αλλά και για να μεταφραστεί σε πρακτικές δράσεις όλη αυτή η ε, θεωρία. Καλωσορίζουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, του σχεδίου δράση. και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σα κάποιε προτάσει και να συζητήσουμε. Κάποια γενικά σχόλια. Είναι υψίστη τη σημασία τα κράτη-μέλη τη Ένωση, να εξασφαλίσουν ότι οι αρχέ που καθορίζονται στον, στην συνένεση είναι, θα γίνουν κατανοητέ και οι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί θα γίνουν πραγματικότητα ε, από τις διάφορε υπηρεσίε, καθώ επίση και από τον στρατό. Πέρα από αυτό, το, ο συμβασμό λέει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εργαλείο διαχείριση κρίσεων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, γιατί μπορεί να έχει επιπτώσει στι ε, ανθρωπιστικέ δράσει τη Ένωση. Οι αποφάσει για την ανθρωπιστική βοήθεια ήταν η απάντηση για τα θύματα της, ε, των καταστροφών. Τώρα έρχομαι στο πρόγραμμα δράσης να σας ε, πω ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να ε, ε, επικεντρωθεί στα βασικά στα εξή θέματα. Ενίσχυση των υποδομών, ενίσχυση των δυνατοτήτων, αντιμετώπιση των, κλιματικών, των κλιματικών αλλαγών, πρόθεση των πολιτικών για την αντιμετώπιση των κρίσεων σε διεθνές επίπεδο και αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών για την ενίσχυση ε, τη δυνατότητα ανταπόκριση. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ να δημιουργήσει μια συνολική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των υποδομών και σε διεθνέ επίπεδο και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι επίση σημαντικό να έχουμε ε, ετοιμότητα για την αντιμετώπιση και αυτό να γίνεται και σε τοπικό επίπεδο. Τα μεγάλα κοινά που υπάρχουν βρίσκονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στι χώρε που πραγματικά χρειάζονται ε, την βοήθεια γιατί αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικέ κρίσει. Η δυνατότητα λοιπόν Λοιπόν αυτή έχει να κάνει με την επένδυση στην, ε, στις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής και έχουμε έτσι καταφέρει ε, να μπορέσουμε να έχουμε ομάδες συντονιστικές, 21 μονάδες ανταπόκρισης με το τεχνικό προσωπικό, πάνω από 180 εκπαιδευμένους εθελοντές έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε έγκαιρα προγράμματα για, τα, για ψυχοκοινωνικά, ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση, ασφάλεια τροφίμων κλπ. Δεύτερον, για τις ανθρωπιστικέ συνέπειε ε, των κλιματικών αλλαγών. Καλωσορίζουμε τις ε, δράσει της Γενικής Διεύθυνση ΕΚΟ για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ε, τονίζει τις ανθρωπιστικές συνέπειες και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω πολιτικών δράσεων για την ανακούφιση και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, καθώ επίση και με την υποστήριξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Η, η συνένεση εκφράζει την ε, ε, επιθυμία να αντιμετωπιστούν όλα αυτά μέσω ε, νομοθεσίας και δράσεων και να βελτιωθεί η κατανόηση των κρατών μελών για όλα αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι οργανισμοί αναγνωρίζουν την συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ για την χρήση των κατευθυντηρίων γραμμών. Το χρηματοδοτικό μέσο του 2009 για την ε, αντιμετώπιση των κρίσεων και επίσης συστήνουμε η αναθεώρηση των, ε, του σχεδίου δράσης να περιλαμβάνει τα εξή. Τα θεσμικά όργανα, ειδικά η Γενική Διεύθυνση για τις Εξωτερικές Σχέσεις, Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Ανάπτυξη, θα πρέπει να ευστήσει την προσοχή της στις κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν μεταξύ για το διάλογο που υπάρχει μεταξύ των μελών που λαμβάνουν τη βοήθεια αυτή και επίσης θα πρέπει να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των ε, κρατών μελών που ε, βασίζουν τις ε, προσπάθειές τους στις κατευθυντήρες αυτές γραμμές και θα πρέπει να ενισχυθεί η διάδραση και με δυνατότητα εξωτερικής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών. Τώρα, για την, για την ανθρωπιστική βοήθεια είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τι ανθρωπιστικέ που υπάρχουν. Επίσης, εναρμόνιση όσων ε, αντιμετωπίζουν αυτές τις ε, διαδικασίες. Πρέπει να είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες αυτές, ειδικά σε ό,τι αφορά το LRD. Θα πρέπει να ε, συνεχιστεί η ενίσχυση των όσων βρουν σε ανθρωπιστικό επίπεδο στις χώρες αυτές. Πρέπει να είναι σαφή, σαφώς καθορισμένα και να γίνονται σεβαστά τα καθήκοντα και η εντολή που έχουν οι άνθρωποι αυτοί όταν δρούν. Ευχαριστώ. Merci. La parole est maintenant au... Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν ε, οι κύριοι βουλευτές. Ο κύριος ε, Γκέρενς έχει ζητήσει το λόγο. Μέχρι να τον περιμένουμε, να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενσολό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Επιτροπή και τους εκπροσώπους των όργανων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήραν το λόγο. Ε, εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια καλή χρονική στιγμή για να προωθήσουμε την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε μια γενική συμφωνία για τη συνένεση που επετεύχθη το 2005 και έχουμε, όπως υπογνωμίστηκε, και μία επίτροπο η οποία ακριβώς έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ανθρωπικής βοήθειας και την ε, διαχείριση κρίσεων, την απάντηση της κρίσης και πρέπει να αναθεωρήσουμε και το σχέδιο δράσης μας ε, να προβούμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, κάνει αυτό που μας ζήτησε ο κύριος Σίγκελ, ε, δηλαδή ε, να σας υποστηρίξουμε στην εκπόνηση της νομοθεσίας, ε, στην εξέβριση των πόρων ε, και στο διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τους εθνικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι εκπρόσωπος της Voice μας ε, αναφέρει το εξής. Ε, εδώ δεν θέλουμε να εοποιήσουμε όλες τις δράσεις ε, των διάφορων οργανισμών που είναι συμπληρωματικές, αλλά σίγουρα θα ήταν καλό να έχουμε καλύτερο συντονισμό και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της αναθεώρησης για να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις των ανθρωπιστικών οργανισμών των κρατών μελών με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συντονίσουμε επίσης καλύτερα τη δράση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δράση άλλων διεθνών οργανισμών, κυρίως με τα Ηνωμένα Έθνη και επίσης να συντονίσουμε καλύτερα την δράση της ε, ε, απάντησης, ε, της ανταπόκρισης που έχουμε σε περίπτωση κρίσεων έτσι ώστε να δίνουμε και ανθρωπιστική απάντηση αλλά και στρατιωτική απάντηση. Στις παρεμβάσεις ακούστηκαν δύο δεινά που θέλω να υπογραμμίσω. Καταρχήν, να μην ξεχάσουμε τις κρίσεις που υπάρχουν παγκοσμίω και που δεν εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε δραματικέ στιγμές. Δηλαδή, να μην διατρέχουμε το κίνδυνο να συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το ενδιαφέρον των ε, ΜΜΕ για να ανταποκριθούμε σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Γιατί, ωραία, προφανώς η IT, στην IT υπήρξε μια δραματική και θεματική καταστροφή, αλλά υπάρχουν και άλλες κρίσεις στον κόσμο που δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε γιατί θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε αυτά που κάθε στιγμή προσελκύουν την προσοχή μας και επιζητούν την προσοχή μας και επίσης ε, να ε, φροντίσουμε να έχουμε μηχανισμούς πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης. Και θα ήθελα να ρωτήσω την ε, Επιτροπή πώς προχωρούν η πρωτοβουλία λόγου χάρη της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Παρέμβασης Πρόκειται για ένα σώμα που θα μπορούσε να παρεμβαίνει σημαντικά σε περίπτωση κρίσης. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέρεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πατήσω φορό τιμή σε, σε όλους όσους είναι παρόντες ε, εδώ με τις ιδιαιτερότητές τους. Ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, ε, το έγγραφο της Συνένεσης ε, αναφέρει πράγματα με τα οποία όλοι συμφωνούν, όμως ε, υποθέτω ότι υπάρχουν και διαφωνίες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ενδεχόμενες διαφωνίες ή σε δυσκολία συμφωνία συμφωνίας ορισμένες πτυχές. Θα ξεκινήσω από την αρχή της αμεροληψίας. Κατά την άποψή μου, δεν ε, ορίζεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρουμε συγκεκριμένα στο MSF. Δεν ξέρω αν ε, η MSF εκπροσωπείται από τη Voice, ε, αλλά η MSF, παραδείγματος χάρη, αρνείται τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες όπου υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Ήταν η περίπτωση του Κωσυφοπεδίου ήταν και περίπτωση, είναι και περίπτωση του Αφγανιστάν σήμερα, ενώ άλλες οργανώσεις όπως η Καριτάς, η DCCR, η Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, έχουν λιγότερο αυστηρά κριτήρια ως προς την εφαρμογή του κριτηρίου της αμεροληψίας. Ε, υπάρχει ε, υπάρχουν εδώ αυτές ε, οι διαφορές, εξακολουθούν να παραμένουν ή υπάρχει μια προσέγγιση. Πρέπει να το δούμε αυτό. Επίσης ε, θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της μεροληψίας. Υπάρχουν καταστάσεις που συγκρούονται μεταξύ τους ή υπάρχουν και διάφορες περιπτώσεις που ακόμα και αν είμαστε μερόληπτοι είναι δύσκολο να δράσουμε. Σκεφτείτε τη Βερμανία πριν κάποια χρόνια είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις, ε, όμως ε, είδαμε ότι, κάποια, ότι η χώρα αυτή είχε κλείσει τα σύνορά της, ε, ακόμη και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση για το Γραφείο Συντονισμού της Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Εγώ θεωρώ και πολύ νομίζω το βλέπουμε έτσι, ότι η κυρία Γεωργίευα έχει την πολιτική ευθύνη στον τομέα αυτό. Αυτή είναι η οποία μπορεί να εγγυηθεί το σεβασμό της αρχής της αμεροληψίας. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται ε, να σκεφτούμε κάτι παραπάνω πέρα από τα κίνητρα ε, για να χορηγήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Όλα αυτά δεν τα λέω για να σας δυσκολέψω, αλλά για να σας παρουσιάσω πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση. Αν στην περίπτωση της Βρεμανίας, ε, λόγου χάρη, ε, δεν βλέπετε την, τον διαχωρισμό ε, το, ε, των ατόμων που εργάζονται στο θέμα αυτό. Καταρχήν, η κυρία Στον δεν μπορούσε να ανοίξει τα σύνορα και να προσπαθήσει να πείσει ε, τους αρμοδίους να ανοίξουν τα σύνορα ε, και κατόπιν οι αρμόδιοι εργαζόμενοι να μπορέσουν αμερόληπτα να δράσουν. Νομίζω ότι κανείς δεν τον αμφισβητεί εδώ αυτό στην αίθουσα και θα πρέπει να δούμε αν κάτι τέτοιο χέρι συνένεσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέβα. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους τα τελευταία 50-60 χρόνια δουλεύουν πολύ σκληρά ε, για τα ζητήματα τα ανθρωπιστικά, για να βοηθήσουν τον κόσμο να ανακάμψει από σοβαρές καταστροφές και έχουμε εδώ εκπροσώπους ε, οργανισμών ε, που είναι πραγματικά εξαιρετική. Εγώ ήμουν στο τσουνάμι στη Σρι Λάνκα όταν έγινε. Πέντε ακροάσεις έγιναν στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει ο κόσμος να ανακάμψει και να επανέλθει στην κανονική του ζωή μετά από το τσουνάμι και άκουσα τα σχόλια του Προέδρου της Σρι για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα πράγματα και άκουσα επίσης ε, και τι υπόθηκε για το Αφγανιστάν και για το Κονγκό. Υπάρχει μια εντύπωση ότι κάποιοι από τους παίκτες ε, στα ζητήματα τα ανθρωπιστικά δεν λαμβάνουν ε, το, το σεβασμό που θα έπρεπε. Μου είπαν, πηγαίνετε σε όλα τα πολυτελή ξενοδοχεία και θα δείτε. Είναι γεμάτη από ανθρώπους ε, της διεθνούς κοινότητας Μάλιστα κάποιος μου είπε εγώ δεν θέλω άλλους μπλιμπάν στη χώρα μου. Τι θέλω να πω. Πώς 136.000 ε, άνθρωποι να γυρίσουν ε, στην ε, χώρα τους. Τέσσερα χρόνια χρειάστηκε αυτό στη Σρι 2,2 δις όμως υπάρχουν στο καταπίστευμα και δεν χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται επί τόπου δεν είναι λεπτομέρεια. Και το λέω αυτό γιατί είναι αντίδραση των χωρών που είναι αποδέκτες της βοήθειας αυτής. Ότι έρχονται διεθνείς διάφοροι, πηγαίνουν σε μεγάλα και πολυτελή ξενοδοχεία, ε, ξοδεύουν λεφτά κλπ. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται και δεν φτάνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς μετά το τσουνάμι δεν θέλει κανένας πλέον η διεθνή κοινότητα στην Ινδία να, να έρθει να βοηθήσει την κατάσταση. Oui, Madame vous avez la parole. Oui, j'aurais voulu savoir. Ναι. Σε σχέση με το εθελοντικό σώμα, θα, θέλα, θα θέλαμε να μάθουμε σε σχέση με τους ε, παραδοσιακούς ε, εταίρους ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια, ε, πώς ε, ακριβώς θα δρουν. Το έχετε σκεφτεί? Ο κύριος Βάγκελ. Ένα ερώτημα θέλω να θέξω σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε να έχουμε έτσι μια συνεκτική πληροφόρηση για το ποιες είναι οι συνθήκες της προσβασιμότητας στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια και ποια είναι τα προβλήματα. Δεν θα έβλαπτε νομίζω την ε, αμεροληψία σας εάν εσείς ή κάποιος από τους οργανισμούς σας μπορούσατε να συμβάλλετε ε, σε τέτοιου είδους πληροφόρηση. Συνέχεια μιλούμε για την κατάσταση στη Γάζα, αλλά υπάρχουν και άλλες παρόμοιες καταστάσεις αλλού, όπου οι πληροφορίες για τις συνθήκες και πώς μπορεί δηλαδή η ε, ε, βοήθεια να φτάσει αυτούς που τη χρειάζονται, οι συνθήκες είναι πολύ εύθραυστες και περίπλοκες. Οπότε χρειαζόμαστε αυτή την πληροφόρηση, χρειαζόμαστε την κειμενική πληροφόρηση. Όχι δηλαδή, όχι για να βασιζόμαστε στην κυβερνητική προπαγάνδα ή στην προπαγάνδα της αντιπολίτευσης ή στην προπαγάνδα οποιοδήποτε, ε- οποιοδήποτε έχει συμφέρον να πει κάτι συγκεκριμένο για την κατάσταση αυτή. Εμείς θα θέλαμε τις δικές σας πληροφορίες. Είναι μια ιδέα... Ίσως θα μπορούσε κάποιος τρόπος να βρεθεί για να καταλήξουμε σε, αυτή την, ε, σε αυτό το χρήσιμο και αντικειμενικό εργαλείο που χρειαζόμαστε στη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στρίφλα, έχετε ζητήσει το λόγο. Ναι, κοιτάξτε. Η Ευρωπαϊκή Συνένεση εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράση από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ε, Δυστυχώ ε, παρέμεινε νεκρό γράμμα στα κράτη-μέλη. Εγώ έχω σκοπό να το παρουσιάσω στην ε, ε Γαλλική Εθνοσυνέλευση, αλλά κατά τα υπόλοιπα δεν έχει προχωρήσει πολύ. Έχουν τώρα το λόγο οι ομιλητέ για να απαντήσουν στα ερωτήματα που του ετέθησαν από του Ευρωβουλευτέ. Ποιο θέλει να ξεκινήσει. Euh, Κύριε Γενική Διευθυντή, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις ε, και σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. και σας ευχαριστώ πραγματικά γιατί στο παρελθόν δεν ε, λάβαμε ιδιαίτερη ε, προσοχή και χαίρομαι ιδιαίτερα για τις παρατηρήσεις ε, που ακούσαμε τελευταίως και στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και επειδή έχουμε πλέον ένα επίτροπο, μία επίτροπο για την ανθρωπιστική βοήθεια, όλα αυτά τα ζητήματα πραγματικά ενισχύουν ε, τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως ακριβώς δείχνουν και οι δύσκολες ερωτήσεις ε, που μου ετέθησαν. Θα ήθελα να σας πω μία ιστορία. Όταν ακούσαμε ότι θα υπάρχει επίτροπος για τα για ανθρωπιστικά ζητήματα συγκεκριμένα, πραγματικά φάνηκε κάποιος ε, ενθουσιασμός. Νομίζω ότι όλοι μας ε, ε, όλοι μας χαρήκαμε, γιατί το γεγονός ότι πλέον η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι υπό την, το ευρύτερο θέμα της διεθνούς συνεργασίας, νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ, ειδικότερα στην ΑΕΤ. Στην ΑΕΤ είδαμε καθαρά από τις 13-14 Ιανουαρίου όταν αρχίσαμε σιγά σιγά να εντοπίζουμε τις ε, ανθρωπιστικές παρεμβάσεις που θα έπρεπε να κάνουμε και πώς ακριβώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε ανάγκες της κατάστασης, ε, είναι γεγονός ότι το αναπτυξιακό ζήτημα αναφερόταν πάντα σε όλες τις συζητήσεις και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και μπορεί να μην απαντήσω ξεχωριστά σε κάθε μία από τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών, αλλά είναι γεγονός ότι έχει να κάνει και με την προετοιμασία για την ε, διάσκεψη για την ΑΕΤ που θα γίνει σε 15 μέρες στη Νέα Υόρκη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν τη διάσκεψη να ασχοληθούμε, να συλλέξουμε στοιχεία σε σχέση με τα ποσά που μεσοπρόθεσμα θα διαθέσουν και οι αρχές της ΑΕΤΙΣ για να αντιμετωπίσει την πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει τώρα η χώρα, αλλά είναι επίσης σημαντικό να μάθουμε σύντομα ποια είναι τα αποτέλεσματα των παρεμβάσεων μη ανθρωπιστικού χαρακτήρα. γιατί καταλαβαίνετε ότι για την ανθρωπιστική παρέμβαση εμείς μπορούμε σιγά σιγά να φύγουμε όταν ε, θα αναλάβουν άλλοι. Και δεν το λέω αυτό για εγωιστικούς λόγους, για λόγους συνοχής το λέω. Και επειδή μιλάμε για την IT, είναι τόσο σημαντική η κρίση στην IT που μας απασχολεί όλους και ναι, μεν πρέπει να δώσουμε προσοχή, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και άλλε αιστείε προσοχή ε, που δεν σταμάτησαν να υπάρχουν στι 12 Ιανουαρίου και δεν έχασαν και τη σημασία του επειδή υπήρξε ο σεισμό στην Αϊτή. Και το λέω αυτό απαντώντα σε κάποια από τα σχόλια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην μας διαφεύγει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα μέσο αντίδραση στην κρίση και όχι διαχείριση της κρίσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζουμε. Και νομίζω ότι το υπενθύμησαν ε, κάποιοι από, κάποιος από, το υπενθύμισε κάποιος από τους ομιλητές ε, σήμερα. Και έτσι απαντάω και στην ερώτηση του κυρίου Γκέρενς τι κάνουμε ε, σε μία, στην περίπτωση για παράδειγμα της Βυρμανίας ή της Σρι όταν υπάρχουν σοβαρά πλήγματα και πώς διαχειριζόμαστε τι συνέπειε τη κρίση. Κοιτάξτε, εμεί ε, στην εντολή μας και δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί η έξοδος από την κρίση. Δεν λέω βέβαια ότι μα είναι αδιάφορο αυτό το θέμα ή ότι δεν έχουμε κανένα αντίκτυπο, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε αυτό. Εμεί πάρα πολύ αξιοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε επί τόπου έχουμε τη δυνατότητα πολλές φορές, ε, ε, τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο εμείς σε ορισμένες ζώνες και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε με καλό τρόπο όλες αυτές τις ε, πληροφορίες σε συνεργασία με το Ρέλεξ. Ενδεχομένως η Μιανμάρ να μην είναι η πιο υποσχόμενη περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφόσον καταφέραμε να μπούμε, καταφέραμε να μπούμε επειδή ακριβώς επειδή υπήρχε ε, μια ανθρωπιστική παρουσία εκεί και υπήρξε μια, υπήρχε μια κάποια αξιοπιστία και μια κάποια δυνατότητα πρόσβασης. Ήμασταν γνωστοί δηλαδή ως εταίροι, ενδεχομένως όχι πάρα πολύ ευπρόσδεκτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάναμε μια χρήσιμη δουλειά. Και γι' αυτό μας αποδέχθηκαν. Επίσης ο κύριος Ντέβα έθεσε το θέμα της Σρι που εξακολουθεί να είναι στο πρόγραμμά μας. Γνωρίζουμε ότι, ότι είχε, είχε έρθει και μια σημαντική αντιπροσωπεία εδώ στην αρχή της εβδομάδας και ε, είχα το προνόμιο, την ευκαιρία να του συναντήσω. Υπάρχει λοιπόν μια ανθρωπιστική προσπάθεια με καλό συντονισμό, ε, γενική διεύθυνση ε, μας βοήθησε Περάσαμε και μηνύματα πέρα από τα καθαρά ανθρωπιστικά και από τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούσαν καθαρά τον εμφύλιο πόλεμο. Όταν κάτι δεν μαθαίνεται στον τύπο, όταν δεν το ακούμε, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν πράγματα στη Σρι Λάγκα δεν φτάνουν πάντοτε όλα στα αυτιά των ε, ε, ευρωπαϊκών οργάνων και επανέρχομαι έτσι στο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης και της ε, Επιτρόπου για το ζήτημα αυτό. Έχουμε μια ανεξαρτησία και είμαστε ουδέτεροι για να μπορέσουμε να έχουμε έναν διάλογο ανθρωπιστικό, να μπορούμε να συντονιστούμε με τα άλλα μέλη της οικογένειας Δέλεξ που εξακολουθούν να υφίστανται εκτός από την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να μπορεί να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς όφελος της ανθρωπιστικής δράσης αλλά και των ε, σχέσεων με τους υπολείπους εταίρους. Μιλήσατε για ε, την Γάζα, Η κυρία Γεώργιεβα το έχει και αυτό στι προτεραιότητε τη και το ίδιο ισχύει για το Τσάντ και για πολλές άλλες περιοχές. Δεν θέλω τώρα να σας παρουσιάσω τα πράγματα όλα ρόδινα, αλλά είναι γεγονό ότι υπάρχει συνοχή στην προσπάθειά μας η συνεργασία σας με την Επιτροπή Εξωτερικών Ζητημάτων είναι χρήσιμη. Βεβαίως μπορείτε να γνωστοποιήσετε και την ε, εμπειρία σας ε, και στο Συμβούλιο, είτε στην ε, Κορεπέ, είτε σε άλλα φόρα για να μπορέσουν ακριβώς, να μπορέσουν να γίνουν γνωστότερες οι ανθρωπιστικές μας παρεμβάσεις. Κύριε Γκέρεντς. Ο κύριο Γκέρεν, ε, θέλουμε να δώσουμε καλό νέο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά για να είμαστε πιστικοί για τα μέλη της Επιτροπής εκείνης, θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση. Από ποια στιγμή, από πότε θεωρείτε ότι απειλείται η αμεροληψία σας ε, ως πρωταγωνιστής στον τομέα τον ανθρωπιστικό, δηλαδή σε θεσμικό επίπεδο η Κομισιόν θεωρεί ότι ποια θα ήταν η παρέμβαση που θα μπορούσε να βλάψει την αμεροληψία. Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση χρήσιμη και δύσκολη γιατί προφανώς δεν είναι όλα ιδανικά σε αυτόν τον κόσμο. Ε, δεν μπορώ να σας ε, αφηγηθώ μια ιστορία όπου έχουμε απόλυτη αμεροληψία όμως ε, ίσως ε, θα σας στείλω τις επόμενες μέρες ένα κινούμενο σχέδιο που υπάρχει σε πολλές γλώσσες ε, και εξηγεί το πρόβλημα αυτό. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε λόγω χάρη το πράγμα της IT, αλλά δεν είναι τι, γιατί ε, και αναφερόμαστε σε ένα σενάριο που έχει να κάνει με τρομοκρατία και εκεί αναλύουμε ε, μια ιδανική κατάσταση απάντησης από τους εργαζομένους στον τομέα. Όμως να σας πω ότι εμείς ζητάμε να γίνεται σεβαστή η αρχή της αμεροληψίας, ε, δηλαδή να έχουμε μια παρέμβαση βάσει των αναγκών και η δεύτερη αρχή είναι η εξής. Εμείς ζητούμε από τους εταίρους μας που είναι όλοι ε, εδώ δίπλα μου να διασφαλίσουν και να θέσουν ε, σε εφαρμογή τη διάθεση της βοήθειας. Αυτά είναι πολύ ουσιαστικά, πολύ συχνά. Σε περιοχές κρίσης είχαμε πολύ δύσκολες συζητήσεις όπου υπόθηκε όχι, τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά έτσι, έχουμε ένα αεροδρόμιο και έχουμε ε, και κάποιους ανθρώπους που είναι ε, με χακί και αν τους θέσετε εκεί τότε θα ε, θέσουν ε, στη διάθεση των, των ανθρώπων που τη χρειάζονται τη βοήθεια. όμως πολλές φορές εμείς είπαμε είπαμε όχι, κοιτάξτε είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, το θέμα αυτό και μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπως φαντάζεστε όπου κάποιος μπορεί να πει αν προτιμάτε να πεθάνουν άνθρωποι για να σεβαστείτε το δόγμα σας παρά να αναλάβετε κάποια δράση τελικά δική σας απόφαση πολλές φορές ε, ε, γίνεται η συζήτηση αυτή και η Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού αντιμετωπίζει πολύ πιο συχνά με τέτοια καθημερινότητα. Δεν υπάρχουν όμω τέλειε απαντήσει ε, για την ε, κατάσταση αυτή. Γίνεται μια εκτίμηση του κινδύνου για την δυνατότητα υπεράσπιση των αρχών. Είναι τόσο απλό. Αν θεωρείτε ότι αν κάνετε ε, κάποια αποχώρηση, δεν ε, θα υπάρξει μια βαθμό που θα σας πει. Να μας τα δεις τη δίνα περίπτωση το πράξετε». Πρέπει να σκεφτείτε αν ε, ο αντίκτυπος επί των αρχών θα ήταν τόσο σοβαρός. Και τότε μπορείτε να σκεφτείτε, ναι, θα προσπαθήσω να εξηγήσω, αλλά τελικά δεν μπορώ να το κάνω. Είναι πολύ δύσκολε οι καταστάσει αυτέ και ο καθένα μα ε, πρέπει να κάνει ένα διάλογο με τη συνείδησή του. Είναι μια δουλειά που την κάνουμε κάθε μέρα. Κοιτάξτε, αναφέρθηκα σε αυτό το κόμιξ, γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα που εξηγεί ότι δεν ε, είμαστε δογματικοί επειδή μας αρέσει να είμαστε δογματικοί, αλλά είμαστε δογματικοί γιατί πρέπει στη διάρκεια του χρόνου να ε, διασφαλίσουμε την δυνατότητα πρόσβαση στη βοήθεια όσων έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν ε, δεν θέλουμε να έχουμε ένα δογματισμό απαράδεκτο Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εννοώ. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και το πιο σημαντικό είναι το εξή. Όταν μια κυβέρνηση ρωτά πώ θα παρέμβετε σε ανθρωπιστικό επίπεδο, πρέπει να το εξηγήσετε. Αλλά λέω πάντοτε σε όλε τι προσβετέ που έρχονται στο γραφείο μου για να θέσουν διάφορε ερωτήσει, τους λέω μπορείτε να πείτε από τώρα στον Υπουργό Οικονομικών σας ε, ότι ούτε ένα σέντς, ε, ούτε ένα λεπτό δεν θα στείλει. Γιατί εμείς ε, την υλοποίηση θα την κάνουμε μέσω των εταίρων μας οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και πολλές φορές έχουμε όμως μία δύσκολη αντίδραση από τις αρχές. Συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά και συγγνώμη που μακρηγόρησε, αλλά είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει συχνά. Για να είμαι πλήρης, να προσθέσω μια απάντηση, μάλιστα λέει πρόεδρος, σε ό,τι αφορά τώρα το σώμα των εθελοντών. Θα προβούμε σε μια διαδικασία διαβούλευση ε, τόσο ε, ανοιχτή όσο είχαμε και για το θέμα της συνένεσης. Τέθηκε σε σύγκριση και στη Λισαβόνα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν όμως ε, δύο διευκρινήσεις Όλοι οι αρμόδιοι ε, πρωταγωνιστές ρωτήθηκαν αν ε, η διεθνή αυτή ε, μονάδα θα μπορούσε να σταλεί στην ΑΕΤ και όλοι μου απάντησαν όχι γιατί κοιτάξτε πρόκειται για μια τόσο δύσκολη περίπτωση κρίσης και δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο εκεί νέους εθελοντές. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δούμε ποια είναι η προσθεμένη αξία αυτού του σώματος των εθελοντών, ποια θα είναι τα καθηκοντά τους και πρέπει να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Ζεράρ, θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ. I just want to, ε, to come back to a couple of ε, points that... Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα και ειδικότερα για το ζήτημα της αμεροληψίας, γιατί είναι κάτι το οποίο από ό,τι βλέπω προκαλεί συζήτηση Είμαι, σίγουρη ότι, είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι από την Διεθνή Επιτροπή και από την ε, Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και την Ερυθρά Ημισέλληνο. Κοιτάξτε, οι ενδιασμοί του να ληφθούν ορισμένα κονδύλια από διεθνείς οργανισμούς δεν είναι ζήτημα πολιτικού μέσου ή όχι. Μια διαπραγμάτευση για να έχει κανείς ανθρωπιστική πρόσβαση ή στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής προσέγγισης, μεταξύ των οποίων ε, θα ήταν η διαπραγμάτευση για την ανθρωπιστική βοήθεια και μετά η ύπαρξη ενός πολιτικού διαλόγου, έχει σχέση με το εξής. Κάποιοι δωρητές, ενδεχομένως και κάποιοι Ευρωπαίοι δωρητές, μπορεί να μην είναι υπέρ των επαφών αυτών. Γνωρίζετε αυτήν ε, την επιλογή, την ε, πολιτική της μη επαφής με τη Χαμάς, για παράδειγμα. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται παγίδα τελικά, γιατί προσπαθεί κανείς ε, να προωθήσει αυτήν την ιδέα της αμεροληψίας και μετά οι δωρητές σου λένε να είσαι αμερόληπτο, αλλά από την άλλη δεν ε, θα μα αρέσει και πάρα πολύ να έχει επαφέ με τη χαμά. Οπότε όπω καταλαβαίνετε υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τη ε, διαπραγμάτευση για όλα τα ζητήματα και τη διαπραγμάτευση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Δέβα, ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα πλαίσιο και να εξαρτάται από το πώς έχουν τα, πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να επιτύχει σε ανθρωπιστικό επίπεδο αν δεν λάβει υπόψη του τι συμβαίνει ε, σε επίπεδο ας πούμε πολιτιστικής ευαισθησίας. Ποτέ δεν θα τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο. Η, η προσέγγιση διαπραγμάτευσης στον Ταρφούρ είναι τελείως διαφορετική από ό,τι στο Κονγκό ή σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνει κανείς πάντα υπόψη. Όσον αφορά τώρα την κατανομή των εργασιών, ποιος μπορεί να προωθήσει τι, όπως ε, είπατε, νομίζω ότι στην περίπτωση της ε, βυρμανία η ΑΖΕΑΝ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και εκείνη και πρέπει να τους λάβουμε υπόψη ως περιφερειακούς παίκτες. Εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν είπα ότι βγείτε έξω από τα δικά σας τα τείχη, μιλήστε με άλλους βουλευτές από άλλες περιφερειακές οργανώσεις, ε, ανταλλάξτε απόψεις μαζί τους, για παράδειγμα με τους βουλευτές της Αφρικανικής Ένωσης, γιατί αυτό είναι μια γέφυρα που μπορεί να βοηθήσει εσάς να γνωρίζετε τις ανησυχίες τους και το αντίθετο. Και επίσης κάποια εμπόδια να σταματήσουν εφίστανται. Και επομένως η μελλοντική ε, πρόσβαση θα είναι ευκολότερη. Ο συντονισμός ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ μιλάμε για ανταγωνισμό των ανθρωπιστικών ε, οργανώσεων, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Ο συντονισμός λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό πράγμα. Μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω εγώ ως εξωτερικός παρατηρητής, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως φόρουμ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει ορισμένα ζητήματα και να δει επίσης ε, πώς η αναθεώρηση της ε, συνένεσης μπορεί να, έχει, να δώσει σημαντικότερο ρόλο στην ΚΟΕΦΑ ε, ως ε, μέσο. Έχουμε πολλούς μηχανισμούς συντονισμού αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όχι μόνο στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αλλά και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχει και πολύ συντονισμός μεταξύ της Ότσα και ε, την, ε, τον Τζον Χόλμς ε, και με τον Πίτερ και χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος ε, που η Επίτροπος έχει το χαρτοφυλάκιο για την ανθρωπιστική βοήθεια και θα δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ζήτημα. Θα το, το κάναμε στο πλαίσιο της ΑΕΤΙΣ και θα το, κάν, θα το κάνει φαντάζομαι πολύ περισσότερο. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων λοιπόν και Μπορεί να είναι διαφορετικές οι απόψεις, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι προκύπτει από αυτές τις ε, ε, τη συνεργασία που μπορεί να προκύψει από τις διαφορετικές αυτές απόψει και η διάσταση απόψεων μπορεί να μην είναι επιβλαβή τελικά. Το ένα, ένα ακόμη ζήτημα που θέσατε, ο επαγγελματισμός της ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, Πίτερ, το ανέφερες αυτό ως προς τις ανησυχίες σου για την IT. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να προβληματιστούμε περισσότερο γι' αυτό. Υπάρχει ένα εθελοντικό σώμα στον ΟΗΕ αν υπάρχει πρωτοβουλία από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το συμπληρώνει αυτό και θα βλέπει επίση ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, ποια είναι η προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτό που ήδη υπάρχει. Ε, βέβαια, η Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και φαντάζομαι ότι θα το πούνε και οι συνάδελφοί μου ε, επειδή βασίζονται στον εθελοντισμό για τη δουλειά τους, δεν θα πρέπει να στέλνουμε αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με ε, τη δική τους δουλειά. Δηλαδή να προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε σε τοπικό επίπεδο τον εθελοντισμό και μετά να έρχονται και άλλοι εθελοντές απ' έξω με τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, όπως είπε και ο κύριος Δέβα. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα εχθές την Επίτροπο να επικεντρώνεται σε δύο πτυχές τις οποίες εξέτασε, την ασφάλεια των εθελοντών αυτών, αν υπάρξει τέτοιου είδου εθελοντικό σώμα που θα αναπτυχθεί και ο επαγγελματισμός. Πρέπει λοιπόν μετά να το αναπτύξουμε αυτό. Αν υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού, πρέπει να το εξετάσουμε. Υπάρχουν αξιολογήσει. Θα έπρεπε κάπω ε, να το επεξεργαστούμε. Το να φτιάξουμε ένα καινούριο σώμα μπορεί να μην, να ε, διορθώσει αυτό το πρόβλημα της έλλειψης προβληματισμού, ε, επαγγελματισμού. Πρέπει να προβληματιστούμε λοιπόν περισσότερο και ελπίζουμε ότι θα μα δοθεί η δυνατότητα. Μάλιστα. Μία από τις συνέπειες του να μην καταλαβαίνει κανείς ε, το τι έγινε μετά, την, ε, μετά το τσουνάμι και την αναδιάρθρωση είναι ότι δεν επιτράπει καμία διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση στις ε, ε, κατασκηνώσεις των προσφύγων που είχαν δημιουργηθεί. Το τσουνάμι ξέφυγε από, την, από τον έλεγχο όλων, οπότε ο πρόεδρος στην κυβέρνηση είπε ότι δεν θα μπει κανένας στα, στα βόρεια της χώρας. Εννιά μήνες ήταν οι άνθρωποι εκεί στις σκηνέ και κανένας δεν επιτράπει να πάει εκεί. Υπάρχουν λοιπόν συνέπειες. Πολλές συνέπειες όμως μπορεί να ε, αξιολογηθούν από την κυβέρνηση. Και εδώ μπορεί το κοινοβούλιο σας να παίξει ρόλο να γίνει ε, διάλογος με τους ε, βουλευτές της χώρας αυτής. Και ξέρω ότι κύριε εσείς το κάνετε. Γιατί για να κερδίσουμε αυτή την κοινή ε, κατανόηση της ανταπόκρισης που πρέπει να δοθεί, που είναι βασισμένη στις ανάγκες και όχι στην πολιτική ατζέντα, είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούν να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στις δυνατότητες. Χωρίς όμως να εμποδίζουμε ή ο χωρί αυτό να θεωρείται ότι είναι τμήμα μιας πολιτικής ατζέντα. Εκεί πρέπει να συνεργαστούμε. Και με, την, με συνένεση αυτή νομίζω ότι μπορείτε να ανοίξετε το δρόμο ώστε να υπάρξει αυτή η κοινή θεώρηση των πραγμάτων. Κάποιο από τους υπολείπου ε, ομιλητέ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Σε σχέση και με το συντονισμό, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το εγχείρημα που κάναμε με τα διδάγματα, το οποίο θα ξεκινήσει και μεταξύ των κροταμελών και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να εμπλακούν και οι ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Νομίζω ότι μπορεί να μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές ε, πληροφορίες και από τους ε, ανθρώπους που δρούν ε, επιτόπου, και από πάνω προς τα κάτω. Τώρα, για την ουδετερότητα, την αμεροληψία. Νομίζω ότι όντως είναι σωστό ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τομέα των μη κυβερνητικών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Πολλές απόψεις είναι διαφορετικές για το πόσο μακριά πρέπει να είναι κανείς ή πόσο κοντά στον, ε, στη συμμετοχή του στρατού σε σχέση με τις χώρες που είμαστε παρόντες και το Αφγανιστάν είναι το χειρότερο παράδειγμα εξ όλων αυτών και θα έπρεπε να πω ότι η πλειοψηφία των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πολύ διστακτικέ στο να είναι πολύ κοντά στι στρατιωτικέ δυνάμει, γιατί δίνονται λάθο μηνύματα στην τοπική, στον τοπικό πληθυσμό. Παρόλο που είναι δύσκολο να το αποδείξουμε, είναι και αυτό ένα λόγο που σχετίζεται με την ασφάλεια. Είναι λοιπόν σωστό αυτό που λέμε, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε τη δουλειά που κάνουν ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει για να υπάρξουν περισσότερε κοινέ θέσει. Στο δίκτυο είχαμε μια κοινή θέση σε σχέση με τις ε, σχέσεις ε, με το στρατό από τις 85 μη κυβερνητικέ και είμαστε σε διάλογο με τα θεσμικά όργανα και στα κρατημέλη για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμη υπάρχει πολλής δρόμος για να προχωρήσουμε λόγω ακριβώς των διαφορετικών αντιλήψεων. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων είναι πολιτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο προφανή, πιο διαφανή, πιο ορατή. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρει. Αλλά με βάση και αυτά που υπόθηκαν ήδη, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι η ορατότητα στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να, προσπερνά τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και τώρα έρχομαι στο άλλο σχόλιο που έγινε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πληθυσμούς στα, στα νότια της χώρας. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει ε, ρόλο να παίξει, ποιες είναι οι αποστολές που στέλνετε στις χώρες, πόσο προσοχή μπορείτε να δώσετε στην όλη διαδικασία, ακριβώς λόγω και των διασυνδέσεων που έχετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με το κράτος μέλος. Ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι όσο, υπάρχει, όσο περισσότερη ε, δημόσια πίεση υπάρχει σε ό,τι αφορά τις κυβερνήσεις και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, την παροχή πρόσβασης, και δεν μιλάω μόνο για διεθνεί μη κυβερνητικέ οργανώσει, όπω είπε ο κύριο Ντέβα, το ίδιο ισχύει και για τι εθνικέ μη κυβερνητικέ. Γιατί όπω είδατε στο Σουδάν υπήρχαν ε, μη κυβερνητικέ κυβερνήσει από το Σουδάν. Που και σε αυτέ απαγορεύτηκε να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Για το σώμα των εθελοντών. Είναι πολύ σημαντικό. Τέσσερα θέματα σχετίζονται με αυτό. Μας ανησυχεί πάρα πολύ γιατί το όλο κίνημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων βασίζεται στον εθελοντισμό. Οι μη κυβερνητικέ δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρί την ε, εθελούσια εθελοντική δέσμευση και σε εθνικό επίπεδο των ε, πολιτών και επιτόπου. Πολλοί ε, δουλεύουμε μαζί μέσω των τοπικών εταίρων. Οπότε είναι σημαντικό το εθελοντικό σώμα, το σώμα των εθελοντών, να βασίζεται και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωση σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη προς τις ε, χώρες ε, που αντιμετωπίζουν ε, κρίσει. Το αν θα είναι η Ευρώπη πιο ορατή μέσω αυτού είναι δευτερεύον. Είναι σημαντικό, αλλά είναι δευτερεύον. Κάτι άλλο, η ασφάλεια. Όταν δημιουργήθηκε το, το Σώμα των Εθελοντών, το 2003-2005 έγινε αυτό. Ε, από τότε όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα για τις παρεμβάσεις της ανθρωπιστικής βοήθειας και της υποστήριξης. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει και είναι όλο και πιο δύσκολο να διαχωρίσουμε μεταξύ των φυσικών καταστροφών, όπου ίσως να είναι καταλληλότερο να χρησιμοποιήσουμε τους εθελοντές, και σειράξεων, ε, γιατί πολλές φορές ε, καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Το θέμα λοιπόν αυτό μας ανησυχεί πολύ, γιατί μετά από την πρόσβαση που είναι το πιο σημαντικό για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να μπορούν δηλαδή να κάνουν τη δουλειά, είναι αυτό. Και μιλώ και για διεθνείς και για εθνικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι υπάλληλοι των εθνικών ε, ε, μη κυβερνητικών το πληρώνουν πολλές φορές με τη ζωή τους. Είναι αυτοί που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από ότι οι διεθνείς κυβερνητικές οργανώ, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν το Σώμα Εθελοντών να μην αντικαταστήσει τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι λίγο της μόδας τώρα να μιλούμε για τον ρόλο των εθνικών ε, φορέων, των εθνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται και με την ε, πολιτική προστασία. Αλλά πρέπει να, είμαστε, να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν διαφορε, διαφορές μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής για το πώς δρούν οι εθνικοί φορείς και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και το πώ ε, συνεργάζονται. Και η δημιουργία δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντικό. Επίση, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι το ε, σώμα εθελοντών θα πρέπει να βασίζεται σε υπάρχουσε δομέ. Μην δαπανάτε χρόνο και χρήμα να δημιουργείτε νέε φορεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Με καλύτερο τρόπο απλώ. Με πιο καινοτόμο τρόπο. Με δημιουργικότητα. Αντί να δημιουργούμε πολλούς νέους, πολλές νέες υπηρεσίες που ούτως ή άλλως θα χρειαστεί χρόνος για να δημιουργηθούν, για να συντονιστούν, οπότε ο γενικός συντονισμός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο και από εκεί η χρηματοδότησή τους είναι δύσκολη. Οπότε οι ανάγκες αυξάνονται. Ε, αντί λοιπόν να σκεφτόμαστε κάτι καινούριο, ας χρησιμοποιήσουμε καλύτερο αυτό, καλύτερα αυτό που έχουμε. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Ε, παραμένουν ε, και κάποιοι ακόμη που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Τουσάν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των θεμελιωδών αρχών. Μας ε, είναι, ένα είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί και ο κύριος Γκέρενς είναι θεματοφύλακας αυτών των θεμελιωδών αρχών. Ίσως θα έπρεπε να αναφερθούμε σε αυτές τις συγκεκριμένε αρχές της αμεροληψίας, του εθελοντισμού, της ενότητας, ε, του καθολικού χαρακτήρα και τα κινήματα της Ερυθράς Μισελίνου και του Ερυθρού Σταυρού εργάζονται σεβόμενα αυτές τις αρχές τα τελευταία 45 χρόνια γιατί ε, στη Βιέννη το 1965 διακηρύξαμε αυτές τις αρχές, ο Ερθροσταυρός και η και φυσικά όλοι οι διάφορες συνιστώσεις ε, του Ερθροσταυρού και της Ερυθράς Ελλήνου, δηλαδή και της Επιτροπή και η Ομοσπονδία, σέβονται τις αρχές αυτές. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ στον ορισμό της αρχής της αμεροληψίας. Θα αναφερθώ στο κείμενο που υπάρχει στο καταστατικό του κυρμάτων της Ερθρασιμής Ελλήνου και θεωρηθεί σταυρού ότι δεν ε, γίνεται καμία διάκριση για ε, ούτε φιλετική, ούτε θρησκευτική, ούτε για τα πολιτικές πεπιθήσεις κτλ. Απλώς ε, εμείς ε, ουσιαστικά θέλουμε να παρεμβαίνουμε όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους από τα δεινά. Έτσι λοιπόν ε, η αρχή αυτή μας επιτρέπει να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και εδώ συμπεριλαμβάνονται και στρατιωτικοί που έχουν καταθέσει τα όπλα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ουδετερότητα, πρόκειται για ένα επιχειρησιακό εργαλείο με το οποίο εργάζονται οι συνιστώσεις του κινήματος και φυσικά και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις και εδώ θα αναφερθώ και πάλι στον ορισμό γιατί με την αμεροληψία, την ιδιαιτερότητα και την ανεξαρτησία μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον ανθρωπιστικό χώρο, αν θέλετε, που είναι απαραίτητος ε, για να παράσχουμε βοήθεια. Η ουδετερότητα είναι εξή. Προκειμένου να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη όλων, το κίνημα δεν ε, συμμετέχει στι εχθροπραξίε ε, ούτε σε οποιασδήποτε ιδεολογικέ, πολιτικέ, φιλετικέ ε, διανέξει. Έτσι λοιπόν δεν λαμβάνουμε πολιτικές θέσεις ούτε συμμετέχουμε σε εχθροπροξίες και με το μέσο αυτό, με αυτό το εργαλείο της ιδιαιτερότητας, έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση, πρέπει να πληρούνται φυσικά και οι αλλά αυτό διευκολύνει την πρόσβαση και μία από τις ε, θεμελιώδες ε, αρχές επίσης είναι και η ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία ε, μας επιτρέπει να διατηρεί την αυτονομία μας, είναι να διατηρούμε μια αυτονομία για να μπορούμε να δράσουμε. Έτσι λοιπόν, αν δούμε τους δωρητές της Διεθνής Επιτροπής του Ρυθρού Σταυρού και ευχαριστώ την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για τη βοήθειά τους, γιατί χρηματοδοτούν πάνω από το 45% τον προπολογισμό της Διεθνής Επιτροπής. Μπορεί να μας χρηματοδοτεί και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη, όμως παραμένουμε ανεξάρτητοι. Ελπίζω να ήταν χρήσιμες οι διευκρινήσεις αυτές και φυσικά αν επιθυμείτε μπορώ να σας διανύμω και το έγγραφο με τους ορισμούς των αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως θέλετε να κάνετε μερικές ακόμη παρατηρήσεις, κύριε Κρόνεμπεργκ. Ναι. Δύο σύντομες παρατηρήσεις ε, επειδή εκπροσωπώ 186 κοινωνίες σε όλο τον κόσμο και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της ε, ημισελίνου, Νομίζω ότι η δημιουργία υποδομών είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο σημαντικό να έρχονται ξένοι παράγοντες ε, να παρέχουν βοήθεια, είναι σημαντική η ανάπτυξη υποδομών επιτόπου στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει ένα σαφής στόχος προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς ευχαρίστως τότε να συνεισφέρουμε και να συμμετέχουμε και στην ανταλλαγή απόψεων ε, για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε τη συζήτηση αυτή και να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης θα σας διαβάσω τις αποφάσεις ε, της συνεδρίασης των συντονιστών, τα αποτελέσματα. Θα αρχίσω από τα τελευταία αποτελέσματα, σήμερα δηλαδή το πρωί. Αποφασίσαμε γνωμοδότηση για την έκθεση ε, γνωμοδότησης για τα παράγωγα και τη δώσαμε στους πράσινους. Το ζήτημα της χρηματοδότησης της καινοτόμου για την ανάπτυξη θα το ενσωματώσουμε αυτό το ζήτημα στην προφορική ερώτηση ε, για το ψήφισμα που αποφασίσαμε για ενόψη του, της επόμενης συνεδρίασης G20 στο Τορόντο. Επίσης, ως προς την... Ε, όσον αφορά το πέραν από το PIB, αποφασίσαμε να το δώσουμε στην κυρία Μουσκαρντίνη, όπως επίσης και το γεγονός της ε, ανακούφισης ε, της ρήπανσης στην Αφρική και των παροχημένων σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που η Επιτροπή μας αποφασίσει να κάνει έκθεση για αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα ε, την, εξω, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και την αγανάκτηση που εξέφρασαν πολλοί, ότι παρά το γεγονός ότι ο συντονισμός ε, της ανάπτυξης είναι αντικείμενο, είναι επίκεντρο της συζήτηση, η Επιτροπή μας δεν έχει ακόμη ε, τύχη διαβούλευσης σε σχέση με το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, σε σχέση με το να μην βαθμιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έναν απλό εκτελεστικό φορέα. Επίσης αποφασίσαμε με τον κύριο Κατσμάρεκ να συντάξουμε μια γνωμοδότηση για την αποσαφήνιση της θέσης μας και να καλέσουμε την κυρία Άστον για ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό, όπως επίσης για να ακούσουμε την άποψή της ε, στο, για, τη θέση της ε, ανάπτυξης στο πλαίσιο της, εξωτερικής, υπηρεσίας εξωτερικών ε, δράσεων. Επίσης θελήσαμε να καλέσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών για μια συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά δεν λάβαμε περαιτέρω αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα το αίτημα της Επιτροπής Εξωτερικών επισήμως να συμμετέχει στο δεύτερο πάνελ της Δημόσιας Ακρόασης για την Παλαιστίνη, με τον κύριο Μπλερ δηλαδή, αποφασίστηκε ότι πρώτον διατηρούμε την μορφή της ακρόασης και το πάνελ και δεύτερον ο πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών ε, θα είναι μέλος του πάνελ ε, στη δεύτερη ακρόαση μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και την κυρία Κρετού. Μετά από την παρέμβαση του κυρίου Μπλερ, ε, η, Επιτροπή, της, η, Επιτρο, πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης και Εξωτερικών θα κάνουν κάποιες παρεμβάσεις για να ανοίξει η συζήτηση με τον κύριο Μπλερ και στη συνέχεια στην τελική μορφή της ημερήσιας διάταξης θα αναφέρουμε ότι θα γίνεται και μια δεύτερη, ένα δεύτερο πάνελ με την Επιτροπή Εξωτερικών και όλες οι περαιτέρω διαβουλεύσεις θα γίνουν μέσω γραπτής διαδικασίας. Επίσης, ε, δεν αναφερθήκαμε στις αποφάσεις 20 Δευτέρας Φεβρουαρίου και της 1ης Μαρτίου. 22 Φεβρουαρίου αποφασίσαμε ότι μετά από το ψήφισμα της 9 η Φεβρουαρίου που εγκρίθηκε στην Ολομένεια σε σχέση με τη Συμφωνία Πλαίσιο ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, η Επιτροπή μας ε, έστειλε κάποιες συστάσεις ε, στην διάσκεψη των Προέδρων επιμένοντας να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου βασικό στοιχείο ήταν η θέση της αναπτυξιακής συνεργασίας στην θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και της εξωτερικής υπηρεσίας για την οποία λήφθη απόφαση χωρίς καν ε, να διαβουλευθεί κανείς μαζί μας. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων, αποφασίσαμε να αποστείλουμε μια γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής όσον αφορά τις ε, δυνατότητες εξουσίας νομοθεσίας της Επιτροπής μας, κάτι που συζητήσαμε χτες ε, και για την οποία η έκθεση των νομικών υποθέσεων γνωμοδοτεί. Ε, ορίσαμε τον κύριο Μίτσελ ε, ως μόνιμο εισηγητή για το ζήτημα αυτό και ως μέλος της ομάδας εργασίας ε, που αφορούν συγκεκριμένα τις νομοθετικές εξουσίες. Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, είχε αποφασιστεί να προσκληθεί η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής για ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μας, ε, ακριβώς για τη θέση της ε, ανάπτυξης ε, στο θέμα του χαρτοφυλακίου της ε, ανταλλαγή απόψεων λοιπόν ε, με την κυρία Άστον στις 23 Μαρτίου στην Επιτροπή Εξωτερικών και ζητήσαμε, θέλουμε να ζητήσουμε από την κυρία Άστον να έρθει και στη δική μας Επιτροπή. Περνώ τώρα στο αποτελεσμα της συνεδρίας 1η Μαρτίου. Αποφασίσαμε για τις, τέσσερι πρωτοβουλίας όταν θα έχουμε μία θέση ελεύθερη ε, να ακολουθήσουμε την εξή σειρά. Καταρχήν, αξιολόγηση ενδιάμεση του σχεδίου δράση και τη ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, δεύτερον, care Systems στην Αφρικά, συστήματα υγειονομικά στην Αφρική και προβλέπεται και ανακοίνωση από την Κομισιόν. Ε, τρία, ε, έχουμε τα, τα αποτελέσματα της ανάπτυξης ε, στα υψίπεδα των ε, Ιμαλαίων και στο Θιβέτ και την θέση σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη για να δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την ε, δικαιώματα να καλέσουν μια συνδιάσκεψη στην Κολομβία όμως ε, οι συντονιστές δήλωσαν ε, σύμφωνοι να υπάρξει μια κοινή αντιπροσωπεία στην Παλαιστίνη που θα επιτελείται από εκπροσώπους ε, ΔΕΒΕΦΕΤ και προϋπολογισμού και μια εργασίας για την Παλαιστίνη θα συμμετέχουν κυρίες συμμετέχουν θα έχουμε συμμετοχή μάλλον διάφορων ε, προσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ε, η Επιτροπή της Βραζιλίας ε, θα αποτελεί από δύο μέλη του ΕΛΚ και δύο μέλη του ΑΝΣΤΕ. Επίσης ε, θα έχουμε ε, τις 31 Μαρτίου μια συνδιάσκεψη στη Νέα Υόρκη για την ανοικοδόμηση της ΑΕΤΗΣ. Η ε, συνδιάσκεψη της προηγούμενης επέτρεψε να συσταθεί μια επιτροπή ad hoc τριών μελών. Τα ακόλουθα μέλη γνωρίστηκαν ως υπεύθυνοι για την οργάνωση δημόσιων ακροάσεων που θα οργανώσει το 2010 η επιτροπή μας. Παλαιστίνη, κυρία Κρετή, δύο property ownership, ε, Μίτσελ και Ντέβα, ε, συμφωνία για, τις για την Αλία τρίτον, εγώ και η κυρία Λίβινγκ ε, τέταρτον, αναπτυσσόμενες χώρες, κύριος Μπέρμαν και παιδική εργασία και θα συμμετέχουν ε, στην ακρόση αυτή και Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν να έχουμε κοινή ακρόαση για τις κοινοτόμες μεθόδους χρηματοδότησης με ε, την ΤΕΒΕ και την Ισπανική Προεδρία αποφασίσαμε να δεκτούμε αν ε, συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις ε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη χρηματοδότηση δίνουν σεβαστές. Η Κομισιόν μας υποσχέθηκε να έχουμε μια οργάνωση συζήτησης για το FLEGT και οι συντονιστές δέχτηκαν την πρόταση αυτή. Ο 8, ο κύριος Νιούτον διορίστηκε ως αντικαταστάτης της κυρίας Ζολή στην Πιλωτική Επιτροπή ε, για το διάλογο μεταξύ νομοθετών. Να υπενθυμίσω ότι θα ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση στις 3.30. Έπρεπε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα γιατί ο κύριος Φίμπαλξ μπορεί να παρευρεθεί εδώ από τις 5 και μετά για να συμμετέχει στη συζήτηση για την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν στις 3.30.